σε αυτές η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, ζητούν προστασία από εμά φεύγοντας από αιστείες πολέμου και καταδίωξης μαζί με τα παιδιά τους έχοντας διασχίσει με βάρκες στο Αιγαίο ε, στο έλεος των διακινητών που τους εκμεταλλεύονται. Πολλοί χάνουν τη ζωή τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν στα φορτηγά κάτω από ασφικτικές συνθήκες, πνίγονται στη Μεσόγειο. Κυρίες και κύριοι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη, όλο και περισσότεροι χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο. Εμείς δεν μπορούμε να ε, απομονωθούμε ε, υψώνοντας τύχη στην Ευρώπη. Σας θυμίζω κάτι. Πριν από λίγες μέρες το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος κατέστρεψε στην Παλμύρα ανεπανόρθωτα μεγάλα πολιτιστικά αγαθά. Ξεχάσαμε όμως ότι ο διευθυντής του μουσείου στην Παλμύρα πριν από λίγες εβδομάδες δημόσια αποκεφαλίστηκε από τη συμμορία αυτή των εγκληματιών οι άνθρωποι θέλουν να γλιτώσουν ακριβώς από αυτούς τους εγκληματίες όταν έρχονται σε εμά και δεν μπορούμε εμείς να τους εμποδίζουμε με τύχη. Αυτή την παγκόσμια πρόκληση δεν θα την αντιμετωπίσουμε ούτε με εθνικισμούς ούτε με εθνικά μέτρα. Είναι παγκόσμια η πρόκληση και η απάντηση θα πρέπει να είναι κοινή πολιτική ασύλου και προσφύγων. Η Κομισιόν θα μας παρουσιάσει σχετικά μέτρα και πρόταση για έναν μηχανισμό κατεπίγουσας ανάγκης, έκτακτης ανάγκης για την κατανομή των προσφύγων. Βεβαίως ε, το θέμα που αφορά όλα τα θεσμικά όργανα είναι ποια ένωση θέλουμε. Μια ένωση όλων εναντίον όλων ή μια ένωση της αλληλεγγύης. Το καθήκον μας είναι μεγάλο. Ίσως είναι το, η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή την οποία αντιμετωπίσαμε η πολιτική της γενιάς μας. Το Δουβλίνο 3, το Σέγγεν, τα νούμερα είναι μεγάλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ε, ε, πολλά δεινά και μιλάμε για ανθρώπους. Οι άνθρωποι έρχονται σε εμά γιατί μας πιστεύουν, πιστεύουν στις αξίες μας, αλλά τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων χωρών ε, δημιούργησαν αβεβαιότητα σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτούς που μας κάνουν πολλές ερωτήσεις και να πω ότι βεβαίως κάποιος που μπορεί να είναι επιφυλακτικός δεν είναι κατά των προσφύγων αναγκαστικά. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη μας και τις ανησυχίες των πολιτών μας, γιατί τα προβλήματα είναι ορατά και μεγάλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Ένωσης, τους αμέτρητους πολίτες που πήγαν στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ε, σε χώρους, ε, σε τόπους διακοπών ε, και προσέφεραν βασικά είδη χρήσιμα για τους πρόσφυγες που φάνουν. Αυτή είναι μια εικόνα ανθρωπιάς η οποία γλυκαίνει την φρικτή εικόνα των ε, ε, θανάτων όπως ε, του, ο πνιγμός του μικρού Αϊλάν που θα μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη μας.